Ich öffne die Sitzung. η διάταξη. Έγκριση. τη ημερήσια διάταξη. Αντιρρήσει. Όχι. Τότε συνεχίζουμε στο δεύτερο σημείο. Δεν έχουμε διερμηνία για όλες τις γλώσσες, αλλά για τους παριστάμενους υπάρχει διερμηνία, επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, στο θέμα 3 στο εργαστήρι με θέμα την επιστροφή πολιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους. Το 1993 το Συμβούλιο εξέδωσε οδηγία για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το άδεφο κράτου μέλους. Η οδηγία αυτή είχε ως στόχο να συμβιβάσει την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών με την προστασία των εθνικών πολιτιστικών αγαθών. Αποδείχθηκε όμως στο ενδιάμεσο ότι η οδηγία αυτή δεν ήταν τόσο αποτελεσματική όσο θα μπορούσε ή θα έπρεπε να είναι και γι' το λόγο η Κομισιόν προτείνει μια αναδιατύπωση, δηλαδή μια επεξεργασμένη καινούρια μορφή της παλιάς οδηγίας, στόχος της οποίας είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα. κυρία Βεζιά είναι η συγκήτριά μας και στις 17 Σεπτεμβρίου είχαμε κάνει μια πρώτη συζήτηση για αυτό το θέμα. Σήμερα έχουμε, ε, ένα, έχουμε ένα εργαστήρι για να εξετάσουμε τις νομικές πτυχές της πρότασης της Κομισιόν. Προς υποστήριξή μας έχουμε ε, προσκαλέσει τέσσερις εμπειρογνώμονες, την κυρία Κορνού, Διευθύντρια του Ογεμινέν, από το Ερευνητικό Κέντρο για την Διεθνή Συνεργασία σε ζητήματα δικαίου. CEC IRS. Τυπικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το ακρονομίο. Κύριος Φρέγκο, ε, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου. Καθηγήτρια, με συγχωρείτε, που θα μας παρουσιάσει τις, ε, τα αποτελέσματα ε, μελέτης που διεξήγαγε. Επίσης, έχουμε την κυρία Μαρία Σνάιντερ από την Ιούνι Ντρουά Διεθνές Ινστιτούτο για την Ενοποίηση του Ιδιωτικού Δικαίου, τον κύριο Εντουάρ ε, Μπλονσέ, από την UNESCO. Σας παρακαλούμε να μιλήσετε 10 έως 15 λεπτά, αγαπητοί εμπειρογνώμονες, και στη συνέχεια να απαντήσετε σε ερωτήματα των μελών της Επιτροπής. Πρωτού προχωρήσουμε στη συζήτηση, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε το χρονοδιάγραμμα, να σας υπενθυμίσουμε ότι έχουμε ήδη το χρονοδιάγραμμα. Η κυρία Μπεζιά θα παρουσιάσει τη συμφωνία αυτή στις 17 ε, Δεκεμβρίου και τον Ιανουάριο θα γίνει ψηφοφορία. Θα ήθελα να δώσω τώρα την, ε, ε, το λόγο στην κυρία Βεζιά. Κυρία Βεζιά, θέλετε να μιλήσετε. Όχι. Τότε θα δώσω το λόγο στην κυρία Μαρή Κορνού. Ευχαριστώ. Με τον καθηγητό Μαλαφυγό του Πανεπιστήμιου του Μιλάνου αρχίσαμε να βλέπουμε αυτό το θέμα όσον αφορά το σχέδιο αναμόρφωση τη οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Αρχίσαμε λοιπόν να εξετάζουμε αυτό το θέμα ανάμεσα στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και την προστασία της κληρονομιάς, κυρίως του εθνικού πλούτου. Μας ζήτησαν λοιπόν ιδιαίτερος να δούμε το άρθρο 1 και 9 του σχεδίου αναμόρφωσης, ένα πρώτο άρθρο που αφορά τον ορισμό της περιμέτρου των αγαθών που μπορεί να επιστραφούν και τα οποία θεωρούνται ως ανήκοντα στον εθνικό πλούτο και το θέμα ε, της υποχρέωσης επιστροφής. Αυτά είναι δύο σημαντικά άρθρα σε αυτό το σχέδιο αναμόρφωσης. Ε, σας λέω και πάλι είναι μια προσωρινή διατύπωση. Υπήρχε περιορισμένος χρόνος, γι' αυτό ζητούμε συγγνώμη. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτό το κείμενο είναι ένα ενδιάμεσο, δηλαδή προσωρινό κείμενο. Θα σας μιλήσω για τον ορισμό, για το άρθρο 1 και το πώς θα εξελιχθεί, δηλαδή ο στόχος είναι να μην υπάρχει πλέον το παράρτημα, το οποίο προσαρτάται στον εθνικό πλούτο και η κυρία Φρυγκό θα σας μιλήσει για την υποχρέωση Όσον αφορά τον εθνικό πλούτο, ε, το πρώτο το οποίο μου φαίνεται απαραίτητο είναι να εξηγήσουμε ότι συνδέεται αυτή η οδηγία με μια έννοια του άρθρου 36 της συνθήκης, ένα άρθρο το επιτρέπει στα κράτη-μέλη για λόγους προστασίας του εθνικού πλούτου ε, που έχει καλλιτεχνική, ε, αρχαιολογική ιστορική αξία να επιβάλλουν περιορισμό στην κυκλοφορία των αγαθών, εξαγωγέ και εισαγωγές, δηλαδή και Αυτή η έννοια λοιπόν θα πρέπει προτού να δούμε το θέμα της ε, οδηγίας, ε, ε, δηλαδή να διαγραφεί το παράρτημα. Ήθελα να σας πω αυτή η έννοια της επιμέλειας είναι μια έννοια που εκφράζει μια που έχει σχέση με την κυριαρχία, δεν υπάρχει αυτόνομη έννοια του εθνικού πλούτου, αλλά το άρθρο 36 παραπέμπει, παραπέμπει απλώς και μόνον στα κράτη, τα οποία έχουν ε, τη δυνατότητα να ορίσουν εκείνα τι θεωρούν ως ε, αγαθά που ανήκουν στον εθνικό πλούτο. Αυτό είναι θέμα αρμοδιότητας του κράτους μέλους και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εναρμονίσει κανονιστικές νομοθετικές διατάξεις πολιτιστικής φύσεως. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν αυτή την επιφύλαξη που υπάρχει εδώ. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα ορίσουν, θα καθορίσουν τι ε, θεωρούν ως εθνικό πλούτο υπό την έννοια της εσωτερικής τους νομοθεσίας. Παρ' όλα αυτά όμως, Υπάρχουν ορισμένα κριτήρια αυτής της έννοιας, τι σημαίνει εθνικός πλούτος εν γέννη ε, αφορά ε, αγαθά τα οποία έχουν μείζον ενδιαφέρον. Όχι όλα τα πολιτικά αγαθά. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το επενθύμησε το 1968 σε μια υπόθεση που αφορούσε ένα φόρο που είχε επιβάλει η Ιταλική κυβέρνηση και αφορούσε όλα τα πολιτιστικά αγαθά ε, εξηγώντα ε, τις ε, την εξαίρεση του άρθρου 36 και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανέφερε ότι αυτή η διάταξη αφορούσε όχι όλα τα πολιτικά αγαθά, αλλά ορισμένα εξ αυτών. Η έννοια λοιπόν της σημασίας, ακόμα και αν δεν καθορίζεται εδώ, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της έννοιας του εθνικού πλούτου. Όπως σας έλεγα λοιπόν, είναι μια έννοια η οποία κατεκτήμηση του κράτους μέλους μπορεί να προσδιοριστεί και όσον αφορά την εσωτερική νομοθεσία βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ κρατών μελών τόσο επί της ουσίας, δηλαδή ε, το, την περίμετρο όπως λέμε που αφορά την ε, μείζωνα σημασία και όσον αφορά τον ορισμό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να καθοριστεί αυτή η έννοια. Υπάρχουν ε, διαφορές. Υπάρχουν ορισμένε χώρες ε, που προστατεύουν τον εθνικό πλούτο και επιβάλλουν το πιο υψηλό επίπεδο προστασία του εθνικού πλούτου. Τώρα, ο ορισμός στην οδηγία αφορά, όπως σας είπα, το άρθρο 36 είναι τα αγαθά τα οποία θεωρούνται ότι ανήκουν στον εθνικό πλούτο και αυτή είναι η έννοια κλειδί. Δεν χρειάζεται να δούμε το παράρτημα, πρέπει να δούμε αυτή την έννοια και κατόπιν η οδηγία θα δώσει μια κατηγορία, θα ταξινομήσει όλα αυτά ε, τα αγαθά που ενδεχομένως μπορούν να ανήκουν στον εθνικό πλούτο. Και αυτά τα αγαθά λοιπόν ε, θα έχουν ένα επίπεδο αρχαιότητας και ένα επίπεδο αξίας. Τώρα, ορισμένα αγαθά υποτίθεται βεβαίω ότι αφορούν στον εθνικό πλούτο, ε, δηλαδή είναι τα αγαθά που ανήκουν σε εθνικές συλλογές ή σε ιδρύματα. Εδώ έχουμε ως βάση αυτή την έννοια κλειδί, τον εθνικό πλούτο, αλλά διαγράφεται το παράρτημα. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι εδώ. Οι κίνδυνοι που αναφέρθηκαν ήδη είναι πολλαπλή. Πρώτος κίνδυνος. Με συγχωρείτε όμως, εδώ πέρα υπάρχει ένα λάθος Δηλαδή για να μην ε, βλάψει κανείς ε, την ε, οδηγία και όχι τη σύμβαση, η πρώτη ιδέα λοιπόν θα διαγραφεί αυτό το παράρτημα, το οποίο όμως μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα του κειμένου. Δεύτερος κίνδυνος, να μην έχει επαρκή εγγύηση για τα άτομα τα οποία μπορούν να εμπλακούν σε μια διαδικασία επιστροφής αγαθών, όπως οι παίκτες στην αγορά, η νομική ασφάλεια και γενικότερα Υπάρχουν συναλλαγές οι οποίες μπορεί να γίνουν πιο εύθραυστες και να δημιουργήσουν ορισμένους κινδύνους για την ευρωπαϊκή αγορά. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ορισμένε εγγυήσει που παρέχονται ουσίας ή διαδικασίας και εγγυήσει τεχνικής και πρακτικής φύσεως. Πρώτη εγγύηση και για αυτό το λόγο ήθελα πάλι να αναφερθώ στο άρθρο 36. Το άρθρο 36 είναι μια εξαίρεση στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας και επικεντρώνεται στα πιο σημαντικά αγαθά. Συνεπώς, τα αγαθά, εδώ μάλλον, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε νομοθεσία που περιορίζει την κυκλοφορία όλων των πολιστικών αγαθών. Υπάρχει εδώ μια απέτηση η οποία μπορεί να ελέγχεται από τους Ευρωπαίους δικαστές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το πρώτο σημαντικό είναι μια διάταξη που υπάρχει από την αρχή που θεσπίστηκαν οι συνθήκες και δεν συζητείται καθόλου η ουσία του άρθρου 36. Δεν θίγεται το 36 και η εφαρμογή αυτού του άρθρου δεν δημιουργεί διαφορές υπήρξε μόνο μία υπόθεση η οποία έμεσα αντιμετωπίζει το θέμα ε, της έννοιας του εθνικού πλούτου. Δεύτερη ιδέα. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι μιλάμε εδώ για αγαθά τα οποία βγήκαν παράνομα από μια χώρα. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή πρόκειται για αγαθά, αντικείμενα, τα οποια βγηκαν παράνομο απο μια χωρα το θεμα αυτο ειναι έφυγαν, δεν ξέρουμε πώς, χωρίς ε, να συνοδεύονται από τις άδειες εξαγωγής, τα πιστοποιητικά που επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία τους. Τρίτη ιδέα, μπορεί να υπάρξει αμφιβήτηση των παικτών που ενέχονται σε αυτή τη διαδικασία της οδηγίας και φυσικά ε, ή από τη σειρά του αυτοί οι παίκτες μπορούν να αμφιβητήσουν την ποιότητα ε, των αγαθών του εθνικού πλούτου. Αναφέρθηκε επίσης στο σύστημα της ενημέρωσης όσον αφορά την κυκλοφορία ε, των πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, η υποχρέωση της κοινοποίηση ε, των εγγράφων ε, στην Επιτροπή. Το σημαντικότερο είναι ο χρήστης να είναι σε θέση να γνωρίζει την νομοθεσία, όχι όσον αφορά κυρίως τον καθορισμό, τον ορισμό του εθνικού πλούτου, αλλά ευρύτερα σχετικά με τον έλεγχο που επιβάλλει α ή β χώρα ως προς την εξαγωγή των πολιτιστικών αγαθών. <clears throat> Όλα τα αγαθά τα οποία υπόκεινται σε έλεγχο δεν ανήκουν στον εθνικό πλούτο. Εδώ θα υπάρξουν πιθανά αγαθά τα οποία μπορούν να ανήκουν στην εθνική κληρονομιά μιας χώρας, στον πλούτο μιας χώρας. Αυτά όσον αφορά την περίμετρο που είπα της οδηγίας, το πλαίσιο της οδηγίας. Αυτά όπως είπαμε είναι αγαθά τα οποία δεν συνοδεύονται από άδεια και έχουν ε, βγει από τη χώρα παράνομα και για αυτό το λόγο θα πρέπει να επιστραφούν στην χώρα από την οποία έφυγαν. Τέλος, υπάρχει μια δράση των κρατών μελών. Τα κράτη μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή ενός ε, αγαθού που βρίσκεται ε, στα χέρια ιδιωτών. Τέλος, όσον αφορά τις εγγύησεις, θέλω πληρώσω αυτή την παρέμβαση, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να καθορίσουν τι σημαίνει εθνικός πλούτος στο εθνικό δίκαιο. Αυτό δεν είναι εύκολο σας μιλούσα για τη διασπορά ε, των νομοθεσιών, της ποικίλη νομοθεσίας, όσον αφορά τη μεθοδολογία και την ουσία. Αυτό είναι μια εθνική αρμοδιότητα. Είναι λοιπόν δύσκολο, ή μάλλον όχι. Ε, ήδη είναι πολύ δύσκολο να καθορίσουν τον εθνικό πλούτο, αλλά εν πάση περιπτώσει, για, ως προς το αποτέλεσμα, δεν είμαι βέβαιη ότι θα καταλήξουμε σε, το πιο καθησυχαστικό για τους χρήστες. Παίρνω την περίπτωση της Γαλλίας. Στη Γαλλία ήμασταν καλά παιδιά, καλοί μαθητές μετά από το 1992 και καθορίσαμε τι σημαίνει εθνικός πλούτος ε, όσον αφορά την εθνική κληρονομιά και είπαμε ότι ο εθνικός πλούτος είναι εκείνο το οποίο ανήκει στη, στα μουσεία, στις εθνικές συλλογές, ε, ιστορικά στοιχεία και τα ιστορικά αρχεία και όλα τα άλλα αγαθά ε, μείζωνο σημασία που αφορούν τον, ε, την εθνική κληρονομιά. Συνεπώ η κατηγορία είναι ευρύτατη και δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια εδώ για του χρήστε με τον ορισμό που έχει δοθεί. Τώρα, για τον εθνικό πλούτο. Πάλι υπάρχουν χώρες ε, που απαριθμούν πολλά αγαθά συγκεκριμένα. Άλλες χώρες όμως έχουν ανοιχτές κατηγορίες και σε αυτό το τομέα είναι δύσκολο να καθορίσουμε ποια είναι αυτά τα αγαθά. Εκεί όπου μπορεί να εξελιχθεί το κείμενο είναι όσον αφορά την ενίσχυση της υποχρέωσης ενημέρωσης των εθνικών νομοθεσιών. Νομίζω το θέμα της ενημέρωσης μπορούμε να το ενισχύσουμε και όχι μόνο υποχρέωση ενημέρωσης για την έννοια του εθνικού πλούτου, αλλά για τις διαδικασίες ελέγχου των μετακινήσεων των αγαθών. Εκεί ακριβώς η αγορά χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Θα έλεγα εδώ, στο πρώτο στάδιο της μελέτης, ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να διαγραφεί το παράρτημα και επειδή αυτό το παράρτημα δεν καθορίζει την περίμετρο, το πλαίσιο των πολιτικών αγαθών, ε, όσον αφορά την αρχαιότητα και την αξία τους, επειδή η βασική έννοια είναι η έννοια του εθνικού πλούτου, επίσης δεν γνωρίζω, δεν είμαι βέβαιη κατά πόσον η παρουσία αυτού του παραρτήματος, δεν είμαι βέβαιη ότι η αποτελεσματικότητα της οδηγίας η μη αποτελεσματικότητα της οδηγίας έχει σχέση με την παρουσία ή την απουσία του παραρτήματος. Αυτό πρέπει να το δούμε νομίζω. Αυτά προς το παρόν. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ορισμένα στοιχεία σε σχέση με το δεύτερο ε, τμήμα της μελέτης, το θέμα δηλαδή της επιμέλειας θα πρέπει να βγάλουμε το παράρτημα όπου, εκεί όπου υπάρχει μία επέκταση, μία προέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, αλλά θα πρέπει να πούμε επίσης ότι η πρόταση αναδιατύπωσης φαίνεται ότι αφορά το ότι η προαπαιτούμενη επιμέλεια θα πρέπει να έχει μεγαλύτερο εύρος από ότι στο παρόν. Εδώ έχετε ορισμένες λέξεις κλειδιά του, της, νέας έκδοσης, της νέας εκδοχής του άρθρου 9, γιατί θα πρέπει ο υπεύθυνο να καταδείξει ότι προέβαλε την δέουσα επιμέλεια και Εάν το εμπλεκόμενο κράτος δεν προβεί στην επιστροφή, αυτό ε, θα πρέπει να οδηγήσει στον ορισμό μιας αποζημίωσης, αλλά το, το βάρος της απόδειξης διέπεται από το κράτος μέλος το οποίο προβάλλει το αίτημα. Εάν δούμε την πρόταση αναδιατύπωσης, εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν νέα στοιχεία. Καταρχήν δεν γίνεται αναπομπή στον εθνικό νόμο σε σχέση με τη φάση των αποδείξεων. Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν ενιαίοι κανόνες σύμφωνα με την πρόταση αναδιατύπωσης το βάρος της απόδειξης ε, προβάλλεται στον ετούντα και εδώ περιορίζουμε και τη διακριτική ευχέρεια του δικαστή. Γιατί αν δείτε το κείμενο του, το παρόν κείμενο, το παρόν άρθρο, βλέπουμε ότι ο δικαστής θα πρέπει να ορίσει μία αποζημίωση που θεωρείται δίκαιη σε κάθε περίπτωση, αν είναι πεπισμένος ότι προέβαλε ο τον, την προαπαιτούμενη επιμέλεια, αλλά υπάρχουν και δύο γραμμές που έχουν διαγραφεί, δηλαδή ο δικαστής θα πρέπει να προβάλλει δίκαιη αποζημίωση ανάλογα με την κάθε περίπτωση υπό τον όρο ότι ο ετών καταδείξει ή αποδείξει ότι προέβαλε την προαπαιτούμενη επιμέλεια. Υπάρχει λοιπόν ένας περιορισμός ως προς τη διακριτική ευχέρεια του δικαστή και θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για την ενιαία εφαρμογή του δικαίου. Δηλαδή δεν λαμβάνουμε υπόψη τα επιμέρους εθνικά δίκαια. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαία εφαρμογή του δικαίου και αυτό θα πρέπει να το δούμε και σε άλλα παραδείγματα. Όταν πρόκειται για το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά την ε, ε, συνεργασία πολιτικών και δικαστικών αρχών. Δηλαδή τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό σε σχέση με την καταβολή αποζημιώσεων και ούτω καθεξής. Δεν είναι η πρώτη περίπτωση δηλαδή που μας απασχολεί. Επίσης δεν υπάρχει κανένας ορισμός στις έννοιας της προαπαιτούμενης επιμέλειας, της δέουσας επιμέλειας. Δηλαδή η αναδιατύπωση ακολουθεί το άρθρο 4.4 της ε, σύμβασης ε, του 95 για να δούμε δηλαδή κατά πόσο ε, υπάρχει δέουσα επιμέλεια θα πρέπει να δούμε κατά πόσο λαμβάνουμε υπόψη μία διαβούλευση για, τον, για την επιστροφή του αγαθού που έχει ε, υπεξαιρεθεί και όλες τις ε, άλλες πληροφορίες και τεκμηρίωση που χρειάζεται έτσι ώστε να γίνει και διαβούλευση με τους κατάλληλους οργανισμούς που θα μπορούσε να αναλάβει οποιοδήποτε υπό παρόμοιες συνθήκες. Ε, θα πρέπει λοιπόν critères Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε κοινά κριτήρια για να δούμε κατά πόσο ο αγοραστής προέβαλε την δέουσα επιμέλεια ή ε, υπάρχει μια γενική εφαρμογή της έννοιας χωρίς έναν καλύτερο ορισμό. Τώρα ως προς την εκτίμηση του κειμένου καθεαυτού. Αναρωτηθήκαμε γιατί υπάρχει αυτή η επιλογή να δοθεί, να μην δοθεί ο ορισμός, γιατί διαγράψαμε το παράρτημα και γιατί μιλάμε για δέουσα επιμέλεια. Πρόκειται για μία επιλογή η οποία συμβαδίζει με συγκεκριμένες ενδείξεις που μας έδωσαν οι, τα εθνικά κράτη-μέλη, οι εθνικές διοικήσεις, με βάση και την έκθεση που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώσαμε πράγματι ότι πάνω το, από το 40% των ε, εθνικών οργανισμών είχαν αποφανθεί υπέρ ε, ενός ε, πιο μεγάλου ρόλου της δέουσας επιμέλειας. Πρόκειται για μία επιλογή η οποία συμβαδίζει με την έκθεση που έχει γίνει για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προέβαλε μία ομάδα εμπειρογνωμών όπου συμμετείχαμε η Μαρή και εγώ. Και τελευταία τώρα παρατήρηση, πώς ορίζεται το κανονιστικό, το ρυθμιστικό πλαίσιο, ποιο είναι δηλαδή το μερίδιο του κανονιστικού πλαισίου μέσα στα πλαίσια της δέουσας επιμέλειας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν εθνικές νομοθεσίες που απέχουν πόρο η μεν από τις δε και ως προς την καλή προέρεση και ως προς την δέουσα επιμέλεια. Υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί και γι' αυτό νομίζω ότι η δέουσα επιμέλεια θα πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο της πρότασης αναδιατύπωσης έτσι ώστε να υπάρξει και η, έννοια της εκτίμησης των ε, περιστάσεων που θα απασχολήσουν τον Εθνικό Δικαστή. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη πρότυπα δυνάμει του άρθρου 7 της ε, Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, της Σύμβασης της Βιέννης δηλαδή, του 80, που θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο διεθνής χαρακτήρας πολίσεων και να υπάρξει ενιαία εφαρμογή της σύμβασης, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη την καλή προαίρεση στις πωλήσει και στο διεθνές εμπόριο. Υπάρχουν λοιπόν ερμηνευτικές πρακτικές τις οποίες λαμβάνουν υπόψη τα εθνικά δικαστήρια. Έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα κοινό κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο μέσα στα πλαίσια των εθνικών ε, δικαιοδοσιών ως προς την ε, απόδοση των ε, αγαθών αυτών στα πλαίσια της οδηγίας και νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και έναν άλλον παράγοντα μέσα στα πλαίσια της πρόληψης, ε, δηλαδή ως προς το διεθνές εμπόριο να υπάρχει ένας μηχανισμός προειδοποίησης διακίνησης ε, πολιτιστικών αγαθών όπου να συνεργάζονται οι τελωνιακές αρχές, οι αστυνομικές αρχές και ούτω καθεξής. διότι όταν μιλάμε για ορισμό των αποζημιώσεων θα πρέπει να ενθαρρύνουμε όλους τους παράγοντες της αγοράς να ορίζουν καλύτερα την προέλευση των αγαθών αυτών. Κάτι το οποίο θα είχε θετικότερη έκβαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστούμε πολύ τους δύο μιλητές. Ο λόγος στην Μαρίνα Σνάιντερ από την ε, Ούνιντρο. UNESCO. Bon, alors, si vous Ωραία, η UNESCO ας ε, λάβει το λόγο πρώτη, εφόσον έτσι αποφασίσατε. Bon. Monsieur, vous l'avez... Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ζητούμε συγγνώμη για αυτή την αλλαγή στην, ε, στον κατάλογο των ομιλητών. Αυτό οφείλεται σε θέμα νομικής λογικής αλλά η σύμβαση της UNESCO ε, υπεγράφει πριν από την, ε, τον Ινδουά. Για αυτό το λόγο παρουσιάζουμε αυτή την, την ομιλία τώρα. Si Αν μου το επιτρέπετε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας, καθώς και τη γραμματεία σας, που μας επιτρέπουν να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο συγκαταλέγεται σε, μία από τις βασικές αποστολές της UNESCO. Εγώ είμαι υπεύθυνο για την καταπολέμηση κατά της κυκλοφορίας των παράνομων αγαθών, κυρίως ε, όσον αφορά τη σύμβαση του 70. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω αυτή τη σύμβαση. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχει 124 χώρες που την έχουν υπογράψει. Η τελευταία χώρα ήταν, είναι η Μιανμάρ τον Οκτώβριο του 2013, πρόσφατα. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είμαστε 23 χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της UNESCO. Στον πίνακα αυτό με κόκκινο βλέπετε όλες τις χώρες που είχαν υπογράψει τη σύμβαση του 70 της, ε, στο πράσινο κύκλο είναι οι χώρες που έχουν υπογράψει και την σύμβαση Νιντρουά που ολοκληρώνει τη Σύμβαση του 70 επάνω σε ορισμένα θέματα τα οποία θα εξηγήσει αργότερα η συνάδελφος κυρία Σνάιντερ. Θα δείτε ότι η Γαλλία και η Ολλανδία ε, αναφέρονται με ένα μικρό S το οποίο σημαίνει ότι υπέγραψαν τη Σύμβαση Νιντρουά όταν ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις. Σήμερα λείπουν πέντε χώρες ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Λετωνία, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα. Σε αυτόν τον κατάλογο λοιπόν δύο χώρες ε, παίρνουν σημαντικό ρόλο ε, στην αγορά τέχνης και η επιθυμία μας είναι να ενταχθούν στις υπόλοιπες χώρες. Η σύμβαση του 70 βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Το υπενθυμίζω, Πρόκειται για την πρώτη διεθνή συνθήκη όσον αφορά την καταπολέμηση ε, της ε, παράνομης κυκλοφορίας και επιστροφής ε, των προστικών αγαθών. Οι συνθήκες που υπήρχαν μέχρι το 70 όσον αφορά τα πολιστικά αγαθά ήταν κυρίως η Σύμβαση της Χάγης του 54 και τα δύο πρωτόκολλα της που αφορούν την προστασία των πολιστικών αγαθών σε περίπτωση ενόπλων σειράξεων. Το 70 όμως οι χώρες ασχολήθηκαν με την παράνομη κυκλοφορία των κινητών αγαθών σε περίοδους ειρήνης και κατέληξαν στο, σε αυτή τη σύμβαση που βασίτησε σε τρεις πυλώνες, προληπτικά μέτρα, μέτρα για την επιστροφή των αγαθών και μέτρα όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία. Όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, οι χώρες που έχουν υπογράψει ε, τη σύμβαση θα πρέπει να έχουν εθνικές υπηρεσίες και να θεσπίσουν εσωτερικές πράξεις όσον αφορά ε, την μεταβίβαση κυριότητας, να συμβάλλουν στην πρόθεση των μουσείων ε, και να φροντίζουν για την προέλευση των αγαθών, να ε, κάνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, να θεσπίσουν κανόνες για τις αγορές, για τους εφόρους μουσείων να εκδίδουν πιστοποιητικά εξαγωγών και να επιβάλλουν κυρώσεις όταν δεν τηρούνται αυτά τα μέτρα. Τα μέτρα που αφορούν την επιστροφή των αγαθών. Αυτά άρχισαν να ισχύουν μετά από την έναρξη ισχύου τη σύμβαση. Είναι ένα κανόνα διεθνού δικαίου που δεν μπορεί να αλλάξει. Η σύμβαση αναφέρεται σε μία ανταμοιβή η οποία θα δοθεί στο άτομο που έχει κάθε λόγο να διατηρεί αυτό το πολιτικό αγαθό, αλλά δεν αναφέρει τις λεπτομέρειες άλλες η σύμβαση. Και το θέμα αυτό μας ενδιαφέρει, διότι η νέα σύμβαση διευκρινίζει αυτό το θυμίο. Τώρα η επιστροφή των πολιτικών αγαθών γίνεται κυρίως μέσω των, της διπλωματικής ε, και πολιτικής οδού μεταξύ των ε, συμβαλωμένων μερών, χωρών και ε, είναι ένας από τους περιορισμούς της σύμβασης θα πρέπει να υπάρχουν στον κατάλογο τα αγαθά αυτά να προέρχονται από μουσείο ή από ένα θρησκευτικό ίδρυμα ή από άλλο οργανισμό ή από ένα μνημείο. Αυτός είναι ένας άλλος περιορισμός. Σε διεθνές επίπεδο ε, ε, ε, το άρθρο 9 είναι πολύ σημαντικό, θα ήθελα να επιστρέψω την προσοχή σα, που επιτρέπει σε ένα κράτο μέλο όταν απειλεί την κληρονομιά του και αναφέρομαι σήμερα στην περίπτωση τη Συρία, αλλά αυτό αφορούσε και το Ιράκ πριν από 10 χρόνια περίπου, τότε μπορούν, μπορεί να ζητηθεί μια συντονισμένη διεθνή προσπάθεια προκειμένου οι συμβαλόμενε χώρε να σταματήσουν αυτή την παράνομη διακίνηση ε, των αγαθών των που προέρχονται από χώρε που απειλούνται από φυσική καταστροφή ή από πόλεμο. Το άρθρο 13 της Σύμβασης αφορά τη διεθνή συνεργασία και απαιτεί ε, τη συνεργασία των αστυνομικών αρχών και άλλων αρμοδίων αρχών. Η UNESCO βρίσκεται στο κέντρο ενός δικτύου συνεργασίας που περιλαμβάνει την Interpol, την Παγκόσμια Οργάνωση Τελωνίων, την ε, UNEDC για την καταπολέμηση οργανώνων εγκλήματο, την UNIDROIT βεβαίω, πολλές άλλε αστυνομίες εκδικευμένε όπως της Γαλλίας, της ε, Ιταλίας, της Ισπανίας, το Διεθνέ Συμβούλιο Μουσείων και πολλού άλλου ειδικού φορεί με του οποίου συνεργαζόμαστε σχεδόν καθημερινά. Και φυσικά οι συμβαλόμενε χώρε, άρθρο 15, παροτρύνονται να συνάπτουν διμερεί συμφωνίε που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του όσον αφορά την καταπολέμηση ε, τη παράνομη κυκλοφορία αγαθών και τη επιστροφή αυτών των αγαθών. Σε διεθνέ επίπεδο μπορούμε να αναφερθούμε στι ΗΠΑ που υπέγραψαν πολλέ διμερεί συμφωνίε με το Περού, το Μεξικό, την Ελλάδα και απεδείξαν πολύ αποτελεσματικέ αυτέ τι συμφωνίε. Τώρα, η καρδιά του θέματο. Η οδηγία 93 7 και οι προτάσει που κάνουμε σχετικά με τις διατάξεις της οδηγία. Θα ήθελα να σας πω εδώ ότι αυτή η οδηγία έχει αντικείμενο την αμοιβαία αναγνώριση των νομοθεσιών των κρατών μελών, αλλά εμείς μέσα από την εφαρμογή της Σύμβασης του 70 επιθυμούμε προσέγγιση ακόμα και εναρμόνιση των νομοθεσιών. Αυτό είναι το αντικείμενο ε, της Σύμβασης Unidroit. Στόχος μας είναι να φτάσουμε να κλείσουμε αυτό το δίκτυο της παρανομίας, να υποφεληθούμε από τα νομικά συστήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη, τα οποία ευνοούν ε, την κυκλοφορία επειδή ε, οι εθνικές νομοθεσίες ε, δεν δίνουν δικαιώματα στον κάτοχο του αντικειμένου. Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένες προσπάθειες που γίνονται και χαιρετίζουμε την επικύρωση ε, της ΕΜΕΣ UNESCO από το Βέλγιο και την Ολλανδία. Το Βέλγιο αναθεωρεί τώρα την ομοθεσία του και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό, γνωρίζοντας το δυναμισμό ε, της ε, βελγικής αγοράς τέχνης. Αναφορικά με το άρθρο 1 της οδηγίας, θα ήθελα να αναφερθώ στο σημείο 1 και 9 το άρθρο 1 και το άρθρο 9 συγκεκριμένα. Το άρθρο 1 τώρα. Μας λέει ότι η νέα πρόταση έχει το πλεονέκτημα ότι διευρύνει το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία σε όλα τα πολιτιστικά αγαθά τα οποία καθορίζονται ω ανήκοντα στον εθνικό πλούτο τη κάθε χώρα. Επιθυμία μα είναι να γίνεται λόγος για πολιτιστικά αγαθά που καθορίζονται και δεν είναι, προσδιορίζονται από τα κράτη-μέλη, αλλά δεν χαρακτηρίζονται ως πολιτικά αγαθά. Με αυτόν τον τρόπο παρεκκλίνουμε σε αυτή τη δυσκολία που έχει σχέση. Pour nous, la nouvelle version a également pour έχουν χαρακτηριστεί ως πολιτιστικά αγαθά. Επίσης υπάρχει ένα σύστημα κατηγοριών πολιτιστικών αγαθών που μπορούν να θεωρηθούν ως εθνικός πλούτος και επιθυμία θα ήταν να παραμείνει το παράρτημα. Να διατηρηθεί το παράρτημα, διότι για μας είναι μια επιπλέον νομική ασφάλεια. Πρότασή μας είναι, στα αγγλικά το βλέπετε και στα γαλλικά υπό την έννοια της ε, οδηγίας αυτής ε, το ε, πολιτιστικό αγαθό είναι ένα αγαθό το οποίο θεωρείται ως αρχαιολογική σημασία, ιστορική σημασία σύμφωνα με την νομοθεσία και τη διοίκηση του άρθρου 36 και επιφέρουμε μια επιπλέον αλλαγή δηλαδή που θα ανήκει είτε σε μία από τις κατηγορίες που ορίζει το παράρτημα είτε στις δημόσιες συλλογές που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των μουσείων, των αρχείων, των βιβλιοθηκών είτε ε, στην εκκλησιαστική περιουσία. Ε, η αυτήν αφορά στις δημόσιες συλλογέ θα πρέπει να διατηρηθεί για να διευκολύνει τα κράτη τα οποία έτσι κι αλλιώ θα πρέπει να κάνουν την απογραφή του εθνικού του πλούτου. Πράγματι είναι προτιμότερο για τα κράτη-μέλη οι δημόσιε συλλογέ να προστατεύονται εξ ολοκλήρου από την οδηγία. Η αναφορά ε, στα θρησκευτικά αγαθά θα πρέπει να παραμείνει δεδομένη τη σημασία που έχει η κυκλοφορία των θρησκευτικών αγαθών που προέρχονται κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη. Εκεί η αγορά έχει εξελιχθεί πολύ. Και όσον αφορά το παράρτημα τώρα, υπάρχει ένα σημείο Β που αναφέρεται στο οικονομικό όριο, το οποίο θα πρέπει πιστεύουμε να διαγραφεί, επειδή αφενός είναι πολύ δύσκολο και στην πράξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί και υπόκειται σε οικονομικές διακυμάνσεις που είναι επιβλαβείς όσον αφορά την νομική ασφάλεια του κειμένου. Τώρα, το δεύτερο σχόλιο μας αφορά το άρθρο 9, κυρίως την παράγραφο 3 του άρθρου 9, Μία από τις προτάσεις αναθεώρησης της οδηγίας είναι να αντιστρέψουμε το βάρος απόδειξης όσον αφορά την καλή πίστη, εναπόκειται στον κάτοχο, ο οποίος ζητεί μια αποζημίωση σε περίπτωση επιστροφής, να αποδείξει ότι δεν είχε γνώση της παράνομης φύσης της, της απόκτησης του αγαθού και συνεπώς ε, δίνουμε μια λύση στο πρόβλημα που υπάρχει, δηλαδή την παραπομπή στην εθνική νομοθεσία, που είναι η λύση που προτείνει η Σύμβαση του 70 και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εδώ είναι ένα κενό το οποίο έχει αντισταθμιστεί με τη Σύμβαση της UNIDROIT. Φαίνεται όμως ότι αυτό το θέμα της αντίστροφης του βάρους απόδειξη αμφισβητείται από ορισμένε χώρε, κυρίω ε, από ορισμένες ε, αγορές τέχνης και εμεί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει αυτός ο κανόνας διότι σε ορισμένες χώρες υπάρχει ο κάτοχος καλής πίστης. Γι' αυτό, ε, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταπολεμήσουμε καλύτερα την παράνομη κυκλοφορία των ε, πολιτιστικών αγαθών. Τώρα, η νέα διατύπωση είναι ε, το άρθρο 4 παράγραφος 4 στη σύμβαση Γιουνιδρουά και προχωράει περισσότερο το σχέδιο με τη φράση της τεκμηρίωσης για την προέλευση του αγαθού ε, και τις άδειε που έχουν χορηγηθεί κτλ. Στην τρίτη παράγραφο πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να αναφερθούμε στην καλή πίστη που παραπέμπει στις εθνικές νομοθεσίες και προτιμούμε μία αναφορά ε, στην δέουσα επιμέλεια. Αυτή είναι λοιπόν η πρότασή μας όσον αφορά την τροποποίηση, ο κάτοχος δεν μπορεί όχι να αναφερθεί στην καλή πίστη, αλλά δεν μπορεί να ζητήσει αποζημίωση εάν δεν έχει ε, ασκήσει τη δέουσα επιμέλεια. Εδώ θα σταματήσω κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε το λόγο και βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ερώτημα. Από την Ούνη του Τρουά. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi effectivement de vous remercier de l'invitation qui a été faite à une... Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι ζητήσατε από την UNIDROIT να παραστεί σε αυτή την ε, συνεδρίαση με σχόλια σε σχέση με το σχέδιο αναδιατυπώσης της παρούσης οδηγίας. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι η UNIDROIT είναι ένας από τους κρίκους της αλυσίδας αυτής, αυτού του μοσαϊκού, που ασχολείται με την πολιτιστική κληρονομιά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ε, συμμετέχοντας ε, στην ε, κατανομή ευθυνών όλων των εμπλεκομένων μερών. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το, το σύνολο αυτό του οπλοστασίου προστασίας. Το σημείο εκκίνησης Με συγχωρείτε, έχω ένα πρόβλημα της τις Mais Δυστυχώς υπάρχει ένα θέμα με τις διαφάνειες. Θα δω πώς... Νομίζω ότι θα μπορέσω να το επιλύσω τάχιστα. Euh, Νομίζω ότι οι συνάδελφοι όλοι διαθέτουν τις διαφάνειες αυτές στο φάκελο. Vous avez raison, Madame Έχετε δίκιο, υπάρχει στους ε, φάκελους η παρουσίαση αυτή, δηλαδή το σημείο εκκίνησης είναι η σύμβαση της UNESCO του 70. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης και στην αναδιατύπωση λαμβάνουμε υπόψη αυτό το σημείο εκκίνησης η σύμβαση του 70 αφορά τη συνεργασία και την πρόληψη και επειδή υπήρχαν ορισμένες αδυναμίες στην αρχική σύμβαση, γι' αυτό η UNIDROIT έδρασε σε αυτό το τομέα, διότι μας ενδιαφέρει το ιδιωτικό δίκαιο το οποίο είναι ελλειπές, διότι η Σύμβαση του 70, όπως και η Οδηγία, ορίστηκαν εκ νέου το 93-95 και ήδη από το 80 ασχοληθήκαμε με αυτό τον εμπλουτισμό. Επειδή και η Οδηγία και η Σύμβαση του 70 χρειάζονται ένα ε, εθνικό νόμο εφαρμογής, Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ενιαίο πλαίσιο από τα κράτη-μέλη. Η UNIDROIT, η οποία έχει έδρα στη Ρώμη με 27 μέλη που συμμετέχουν, έχει σαν στόχο να ορίσει ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και νομοθετημάτων. Αυτό είναι ύψης της σημασίας. Δεν θα επανέλθω στον ορισμό και τη διαφορά μεταξύ σύμβασης UNIDROIT και οδηγίας που δίνει τη δυνατότητα στους ιδιώτες να δράσουν για την ε, απόδοση των πολιτιστικών αγαθών. Ε, λαμβάνει υπόψη λοιπόν δύο διαδικασίες, μία για τις κλοπές και μία άλλη για τις παράνομες εξαγωγές. Υπάρχουν λοιπόν δεν θα ήθελα να επανέλθω επί του μηχανισμού που γνωρίζετε αρκετά καλά. Θα ήθελα να μιλήσω για τα περιθώρια παραγραφής, διότι υπάρχουν σχετικά ε, βραχία διαστήματα παραγραφής και άλλα που διαρκούν περισσότερο. Πρόκειται λοιπόν για έναν καθολικό μηχανισμό και γι' αυτό χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να φτάσουμε στον απότερο στόχο. Θα ήθελα να ξαναδούμε αυτές τις προθεσμίες. Βλέπουμε ότι η σύμβαση της UNIDROIT θα πρέπει να εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη έτσι ώστε σε περίπτωση κλοπής να λάβουν υπόψη το ίδιο πλαίσιο με αυτό που ισχύει στην περίπτωση αυτή ε, τον των ε, μάλλον των πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα εξαχθεί. Δηλαδή την περίπτωση της παράνομης εξαγωγής. Άρα η οδηγία αλλά και η σύμβαση UNIDROIT σχετίζονται με μία διαδικασία αποζημίωσης. Μιλάμε για, την, ε, ε, για τον ορισμό της ε, καλής πίστης αλλά και του βάρους της απόδειξης. Και αυτό το βάρος της απόδειξης βαραίνει τον κάτοχο. Ήδη εξ αρχής θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να οριστεί μία αλυσίδα και ο μόνος που μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία είναι ο κάτοχος. Εάν δείξει την καλή του πίστη, είναι ο μόνος που θα μπορούσε να μην αγοράσει αν είχε κάποια υποψία για την προέλευση. Άρα αυτό φέρει και το βάρος της απόδειξης. Εάν ο κάτοχος τώρα έχει το βάρος της απόδειξης, θα πρέπει να του πούμε τι περιμένουμε από αυτόν. Γι' αυτό στην αναδιατύπωση βλέπουμε ότι το άχθος ή το βάρος απόδειξης βαρύνει τον κάτοχο για να υπάρχει μια πιο ενιαία ερμηνεία από τις δικαστικές αρχές. Για να δούμε πώς ορίζουμε και την αποζημίωση. Όμως θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεχόμενος αγοραστής θα πρέπει να έχει τα στοιχεία στη διάθεσή του για να του πούμε τι πρέπει να κάνει, να δει τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση που ανακύψει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή να μιλήσει για την επιμέλεια κατά τη στιγμή της αγοράς. Θα πρέπει να τον βοηθήσουμε. Τι πρέπει να κάνει. Ο δικαστής θα τον ρωτήσει, αλλά θα πρέπει και ο κάτοχος να ξέρει επίσης τι πρέπει να κάνει. Πρόκειται για το άρθρο 4.4 της Σύμβασης UNIDROIT Η UNIDROIT ανέλαβε αυτή την έρευνα που της ανέθεσε η UNESCO γιατί κατά τη δεκαετία του 60 ήδη είχαμε ορίσει την καλή πίστη και κατά τις αρχές της δεκαετίας του 70 θέλαμε να έχουμε όλα τα στοιχεία για να ορίσουμε την καλή πίστη. Δεν θα ήθελα να επανέλθω σε στοιχεία τα οποία ε, αναφέρονται στη σύμβαση UNIDROIT μπορείτε να δείτε ότι τα δύο κείμενα είναι πανομοιότυπα. Υπάρχει ένα στοιχείο επί του οποίου θα ήθελα να επιμείνω και αφορά τη διαβούλευση των ε, ε, παραπομπή στα αρχεία. Διότι όταν μιλάμε για καλλιτεχνικά έργα, το, 1985 το 85 όταν ενεκρίθη η σύμβαση είχαμε το ε, μητρό της Ίντερπολ, της ΟΣΕΒΕΣΕ στη Γαλλία, αλλά επρόκειτο για Μητρό που δεν ήταν προσβάσιμα στο κοινό. Μετά την σύμβαση UNIDROIT υπάρχουν ε, κώδικες ε, δέουσας επιμέλειες για την UNESCO και υπάρχει και ο κώδικας της e-com για τα μουσεία και άλλους φορείς. Ξέρουμε ότι οι έμποροι δεν χρησιμοποιούν αυτά τα μητρώα. Λένε ότι ακόμα και αν τα χρησιμοποιήσουν δεν υπάρχει πιστοποίηση. Αυτό είναι λάθος, μπορούμε να το ζητήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε αυτά τα στοιχεία έτσι ώστε τα ε, εμπλεκόμενα μέρη να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα μέσα. Διότι όταν μιλάμε για παράνομη απομάκρυνση από το έδαφος και όταν μιλάμε για κλαπέντα, για κλοπημαία, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για πολύ σημαντικά αγαθά τα οποία έχουν κλαπεί πριν. Εάν υπάρχει λοιπόν κλοπή και καταγραφή σε μια τράπεζα δεδομένων αυτής της κλοπής, ξέρουμε πότε βγήκαν παράνομα αυτά τα αγαθά. Πολύ συχνά δεν γίνεται χρήση της οδηγίας γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να ορίσουμε την ημερομηνία εξαγωγής. Εάν όμως υπάρχει ημερομηνία κλοπής στα αρχεία, ξέρουμε ότι οπωσδήποτε η εξαγωγή είναι μεταγενέστερη. θα δείτε στα έγγραφα αυτά ότι υπάρχει μία, ε, μία ειδική ρήτρα αναφοράς και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η οδηγία χρησιμοποιείται από τα κράτη-μέλη. Η σύμβαση της UNITRUA επιτρέπει ακόμα και σε έναν ιδιώτη να απαιτήσει το αγαθό που διέθετε. Πριν από το 2002 υπήρχε ο κανονισμός 1215 ε, του 12 που επιτρέπει σε έναν ιδιώτη να δράσει. Έχω το αγγλικό κείμενο μπροστά μου, δηλαδή τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να δράσουν στην ε, περίπτωση απέτησης, λαμβάνοντας υπόψη με το που βρίσκεται το αγαθό. Πρόκειται λοιπόν για ένα νέο στοιχείο που ορίστηκε μετά το 1995 από τη σύμβαση της UNITRUA, γιατί θα πρέπει να, ε, να αχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι υπεύθυνοι εκεί όπου βρίσκεται το αγαθό έτσι ώστε να ληφθούν και ασφαλιστικά μέτρα. Η σύμβαση της UNIDROIT ισχύει σε 34 κράτη, αλλά θα ήθελα να πω ότι 14 ε, κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη συμμετέχουν. Θα θέλαμε βεβαίως να αυξήσουμε τον αριθμό αυτό, αλλά γνωρίζουμε ότι η Γαλλία και η Ολλανδία είχαν υπογράψει, αλλά επειδή αντέδρασαν οι έμποροι δεν, έγινε, δεν είχε γίνει ακόμα κύρωση και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η αναδιατύπωση θα βοηθήσει τα κράτη αυτά στην κύρωση, διότι σε μία μελέτη αντικτύπου διαφαίνεται ότι αν όλα τα κράτη συμμετείχαν στη σύμβαση της UNITRUA, δεν θα χρειαζόταν οδηγία, διότι τα κράτη θα καλύπτονταν πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σωστά όλα αυτά που ακούσαμε. Ωστόσο, πολλές φορές οι προθέσεις μας ε, με τις, ε, δεν, δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στην ορθότητα. Κυρίες και κύριοι, ποιος ε, θα ήθελε λοιπόν... Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μας κάνετε αυτό το θαυμάσιο δώρο για μια ακόμη φορά. Είναι όμως ένα πικρό δώρο θα έλεγα. Δεν θα έλεγα ότι έχω αρκετή νομική κατάρτιση διότι το... πρέπει κανείς να έχει νομική κατάρτιση να καταλάβει όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει όμως, μιλάμε για αυτή την αναδιατύπωση της οδηγίας. Το πεδίο εφαρμογής μας είναι περιορισμένο. Η οδηγία αφορά την επιστροφή ε, των εθνικών πολιτικών στοιχείων ε, που έχουν ε, φύγει από τη χώρα παράνομα δεν θα δούμε όλα τα νομικά προβλήματα που τίθενται όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά, τις παράνομες εξαγωγές πολιτιστικών αγαθών και δεν θα δούμε και τις διάφορες νομοθεσίες μεταξύ των κρατών μελών. Αλλά πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πρόοδου. Ευθύς εξ αρχής το βασικό πρόβλημα ήταν ο λόγος για τους οποίους διαγράφεται το παράρτημα εξεπλάγιν από μια παρατήρηση της κυρίας Κορνού που μας έλεγε ότι και εκείνη ε, αναρωτιόταν κατά πόσον η αναποτελεσματικότητα της οδηγίας του 1993 οφείλονταν στο παράρτημα αυτό το οποίο αυτό αναφέρει ακριβώς η Επιτροπή. Ομολογώ ότι και εγώ προβληματίζομαι και είμαι διχασμένη ανάμεσα την ανάγκη ε, να τηρήσουμε την αρμόδια των κρατών μελών όσον αφορά τον ορισμό του εθνικού τους πλούτου και το συμφέρον που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνει σε αυτά τα θέματα. Μας λένε ότι ο σκοπός είναι να συντονιστούν οι ενέργειες των κρατών μελών. Όπως έχουν τα πράγματα λοιπόν, η σύνταξη του άρθρου 1 δεν με ικανοποιεί. Όσον αφορά τις νομικές διαδικασίες τώρα, κυρίως για το άρθρο 9, νομίζω ότι προχωρήσαμε αρκετά και τα κράτη-μέλη επίσης προχώρησαν σε σχέση με τη θέση του Συμβουλίου επί του θέματος αυτού. Πιστεύω ότι το θέμα της δέουσας επιμέλειας δεν δημιουργεί πλέον πρόβλημα. Και το βασικό ζητούμενο είναι η αναφορά στην καλή πίστη, διότι δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δύο όροι. Θα ήθελα λοιπόν η UNESCO, επειδή ο εκπρόσωπος UNESCO αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, θα παρακαλούσα λοιπόν την UNESCO να μας διευκρινίσει περισσότερο τη σκέψη του όταν μας λέει ότι θα πρέπει να διαγραφεί αναφορά στην καλή πίστη. Συμφωνώ μαζί του εδώ, αλλά θα ήθελα οι παρόντες και οι παρούσες συνάδελφοι να ενημερωθούν περισσότερο. Και γι' αυτό παρακαλώ τους μεν και τους δε. Αν να μας πούν κατά πόσον πιστεύουν ότι η σύνταξη της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 9, όχι λάθος, ναι, η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 9, ναι, κατά πόσον ανταποκρίνεται, πιστεύουν, στην ανάγκη προσανατολισμού, θα έλεγα, της ε, νομολογίας επ' αυτού. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία μας δίνει αυτό το εδάφιο, το δεύτερο εδάφιο, που ακολουθεί την καλή κατεύθυνση αντιθέτως προς το σύνο του άρθρου. Και θα ήθελα να παρακράσω τον κύριο Φρυγκό κυρίως να μας πει τι εννοεί όταν μας λέει ότι ένα διατύπωση της οδηγίας οδηγεί προς μια ομιμορφία του ευρωπαϊκού δικαίου. Εγώ δεν συμφωνώ. Θα ήθελα να μας διευκρινίσει αυτό που λέει. Διότι αυτά που έλεγε στην αρχή της παρέμβασης και στο τέλος της δεν συμφωνούν απόλυτα. Είναι κάπως αντιφατικά. Γι' αυτό θα ήθελα διευκρινήσεις σχετικά επειδή από ό,τι κατάλαβα αυτά που μας είπε για το άρθρο 9, μας είπε ότι τα στοιχεία του άρθρου 9 ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Να μας εξηγήσει όμως παρακαλώ. Πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 9, με συγχωρείτε που επαναλαμβάνομαι και ίσως είμαι και λίγο απότομη, αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ε, ένα θέμα απλό Βρισκόμαστε σε ένα... Ε, δεν μου έρχεται η λέξη, λέει κυρία. Βρισκόμαστε σε ένα έδαφος, δεν μου έρχεται η λέξη. Όχι τόσο ληστηρό όπως ορισμένοι νομίζουν, διότι εν μεταξύ το δίκαιο έχει εξελιχθεί. Υπάρχουν νομικές πράξεις, νομικά μέσα που επιτρέπουν σε ορισμένους ξύπνιους που είναι οι κύριοι παίκτες της αγοράς τέχνης, ε, να χρησιμοποιήσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Και επαναλαμβάνω ότι ο στόχος αυτής της οδηγίας είναι αρκετά περιορισμένος. Δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε όλο το πρόβλημα ε, των πολιτιστικών αγαθών ε, μέσω αυτής της οδηγίας και της εξαγωγής του σε άλλες χώρες. Πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μια θετική κατεύθυνση ώστε όλα τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να καταβάλουν προσπάθειες συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου χώρας. Και προκειμένου να επικυρωθούν οι διεθνείς πράξεις που έχουν οι χώρες στη διάθεσή τους, μόνο τότε θα δώσουμε την καλύτερη απάντηση στο τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ διότι σε αυτό το τομέα κυρίως και αναφέρομαι ε, στη σύμβαση της UNESCO για την πολιτιστική ποικιλότητα, πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε σημαντικός παράγων για την επικύρωση αυτών των πράξεων. Και εδώ νομίζω ότι ο ρόλος της Εύρωσης μπορεί να είναι πιο δυναμικός από ό,τι μας προτείνεται εδώ. Ευχαριστώ, Μαρή Τερέζ. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Απίστευτο. Δεν ξέρω εάν αυτό οφείλεται στην προοπτική των ευρωεκλογών του 2014. Ίσως είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι ως προς ορισμένα θέματα, ιδιαίτερα όταν τα συζητάμε με τους πολίτες μας. Μας μιλούν για την περιπλοκότητα των κανόνων και κανονισμών και για την ανάγκη εναρμόνισης. Πρόκειται για κάτι το ιδιαίτερα δύσβατο και δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει. Η κυρία Κορνού μίλησε για το ενδεχόμενο επιβολής μέτρων στα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πώς μπορούμε να απλουστεύσουμε. Εγώ χάθηκα σε αυτό τον κικαιώνα τεχνικών προδιαγραφών. Θα ήθελα να πω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο το θέμα είναι ιδιαίτερα ε, σημαντικό παρόλο που από εθνικής πλευράς είναι δύσβατο. Θα πρέπει να φτάσουμε σε μια ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσα από τις εθνικές ταυτότητες και την εθνική κληρονομιά, την ε, ταυτότητα των πολιτών και να δούμε τους σημαντικούς αυτούς άξονες που είναι ύψης της σημασίας. Να δούμε λοιπόν αυτή την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά που μας απασχόλησε εδώ και αρκετά χρόνια η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά είναι το συμπίλημα των εθνικών ε, πολιτιστικών κληρονομιών. Θα πρέπει να έχουμε κοινούς, ε, έναν κοινό τρόπο συνδιαλλαγής, ε, συνομιλίας, ιδιαίτερα σε περίπτωση κλοπής αγαθών πέρα από το κρατικό επίπεδο υπάρχει και το περιφερειακό ή στη δική μου περίπτωση ο πολιτισμός της Καταλωνίας και της ε, περιοχής της Οξιτάν είναι ύψης της σημασίας γιατί υπάρχουν και ιδιωτικές συλλογές, όχι μόνο δημόσιες. Θα πρέπει λοιπόν να καταγραφούν όλα αυτά τα συστήματα για να προσπαθήσουμε να συνοδεύσουμε τα κράτη με πιο απλουστευμένα συστήματα από τα υπάρχοντα. Άρα με την αναθεώρηση μιας οδηγίας θα πρέπει να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να απλουστεύσει και να βοηθήσει έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να είναι αποδοτικά σε επίποδο έρευνας, ταύτισης αλλά και κυρώσεων. Ευχαριστώ. Merci bien. Νομίζω ότι η συζήτηση αφορά μόνο Γάλλους ή Γαλλόφωνους. Η γαλλοφωνους κυρια Ραπ... Ευχαριστώ. Δεν θέλω να επανέλθω στο θέμα ότι το το ζήτημα είναι περίπλοκο αλλά και πολύ ενδιαφέρον. Ε, συγκρατώ τρία σημεία. Ακόμα δεν μπορώ να αποφασίσω, χρειάζομαι χρόνο, να αποφασίσω κατά πόσο είμαι υπέρ ή κατά τη διαγραφή του παραρτήματο. Άκουσα επιχειρήματα υπέρ, επιχειρήματα κατά. Είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει σε κρεμότητα και στο δικό μου το μυαλό. Τώρα, όσον αφορά την έννοια της καλής πίστης. Άκουσα ότι η έννοια της δέουσας επιμέλειας είναι μια έννοια που εξαρτάται από τις διάφορες χώρες και η έννοια της καλής πίστης θα ήταν προτιμότερη. Το αντίθετο συμβαίνει. Α, δεν κατάλαβα λοιπόν. Το αντίθετο. Τότε, η καλή πίστη. Λοιπόν, η δέουσα επιμέλεια έχει περισσότερους υποστηρικτές. Πολύ καλά. Το τελευταίο το οποίο μου φαίνεται σημαντικό είναι η υπογραφή και επικύρωση από όλα τα κράτη-μέλη τη σύμβασης ε, της UNESCO. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη σε αυτή την πρόταση ε, για διατύπωσης οδηγίας. Θα μπορούσαμε ίσως κάπως να το εξηγήσουμε ότι είναι απέτηση όλα τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν τη σύμβαση της UNESCO. Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν μια πρόοδος. Ευχαριστώ. Ομολογώ, ευχαριστώ πολύ. Ομολογώ ότι και εγώ δεν ε, καταλαβαίνω πολύ καλά την έννοια της καλής πίστης. Δεν είμαι νομικός. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να το ε, ορίσουμε σε νομική πράξη ε, αυτή την έννοια της καλής πίστης. Νομίζω ότι η επιμέλεια είναι κάτι διαφορετικό. Ορίζεται θαυμάσια. Τι σημαίνει δηλαδή να χειρίζεται κανείς την υπόθεση την εκάστοτε υπόθεση με επιμέλεια. Το πρόβλημα βεβαίως είναι ότι αν δεν ε, επιογράψουν όλα τα κράτη-μέλη, τότε τίθεται το ερώτημα αν, ε, αν υπάρξει οδηγία, τότε ε, δεσμεύει τους πάντες. Από αυτή την άποψη λοιπόν θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε ένα δίλημα. Αν υπάρχουν κάποιες χώρες που δεν θέλουν να συμμετάσχουν τότε δεν πρόκειται να αναδιατυπωθεί και η οδηγία, θα παραμείνει σε ισχύ η παλιά και γι' αυτό αναρωτιέμαι ή μήπως το κατάλαβα λάθος. Αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να ε, λύσουμε αυτό το πολύ δύσκολο πρόβλημα. Κυρία Παδατού, έχετε ένα, ένα ερώτημα. Αυτό το οποίο θα ήθελα είναι ότι στην οδηγία η μηπως το καταλαβα λαθος αναρωτιεμαι πως μπορουμε να λυσουμε αυτο το πολυ δυσκολο προβλημα κυρια παδατου έχει ενα ενα ερωτημα αυτο το οποιο θα υπάρξει αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να περιληφθεί στην οδηγία υπογραφή της σήμερα UNESCO. Αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει κάποιος από την Επιτροπή εδώ? Όχι κανείς και όμως. Αλλά δεν είσαστε ο αρμόδιος επί του θέματος. Εντάξει, πολύ καλά. Ποιος θέλει λοιπόν να απαντήσει. Κυρία Σνάιντερ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα απαντήσω στις ερωτήσεις κύριε Σερζέκ που έκανε αυτές τι ερωτήσεις, αλλά για την δέουσα επιμέλεια και την καλή πίστη τώρα. Δεν θα επισέλθουμε σε όλε τι λεπτομέρειε των διαφορών που υπάρχουν. Σε εθνικό επίπεδο μπορεί να υπάρξει διαφορά. Σε διεθνέ επίπεδο όμω, και οι δύο εκφράσει χρησιμοποιούνται από την ε, σύναψη της UNIDROIT το 1995, εκουσίως επιλέξαμε να αποστασιοποιηθούμε από αυτές τις λέξεις καλή πίστη. Γιατί, επειδή καλή πίστη σε, εθνικό δίκαιο είναι μια πολύ ισχυρή έννοια και ανάλογα με τις περιπτώσεις οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Για παράδειγμα, η προστασία σε αυτό το τομέα, καλή πίστη. Μπορούμε να φτάσουμε στα άκρα. Λοιπόν, για να αποφύγουμε ο δικαστής να μην δεσμεύεται ε, όσον αφορά την εθνική ερμηνεία και τους κανόνες είπαμε ότι αυτό το οποίο ζητούμε είναι μια συμπεριφορά το οποίο ονομάζουμε δέουσα επιμέλεια. Συνεπώς όλοι οι κώδικες δεοντολογίας έχουν σχέση με αυτό. Νομίζω ότι δεν πρέπει ε, σε διεθνές επίπεδο να χρησιμοποιούμε έννοιες όπως η καλή πίστη, το πιστεύω. Δεύτερη παρατήρηση. Η πρόταση να γίνει μια σύσταση στα κράτη-μέλη να προσχωρήσουν ε, στη Σύμβαση του 70. Σίγουρα, γενικά για την προστασία της κληρονομιάς, η Σύμβαση του 70 είναι η αναφορά, το σημείο αναφοράς. Αλλά επί του συγκεκριμένου θέματος επιστροφή των πολιτικών αγαθών και Γι' αυτό πρόκειται εδώ, επειδή η ίδια η UNESCO στη δεκαετία του 80 αντελήφθη ότι η σύμβαση δεν ήταν αποτελεσματική, επειδή παρέπεμπε πολύ στις εθνικές νομοθεσίες και συνεπώς στις διαφορές που υπήρχαν και ζήτησε στην UNIDROIT να καταρτήσει ένα κείμενο το οποίο θα μπορούσε να είναι πρωτόκολλο στη σύμβαση UNESCO, αλλά αποφάσισαν, επειδή εμεί έχουμε ε, στο ιδιωτικό δίκαιο και την εμπειρία και την εντολή, να δημιουργηθεί αυτή η σύμβαση τη UNIDROIT. Και οι μελέτες επιπτώσεων αναφέρουν όχι μόνο ότι αν τα κράτη-μέλη ε, τη Ένωση προσχωρούσαν στην UNIDROIT, τότε δεν είχαμε ανάγκη την οδηγία, αλλά αναφέρει επίση αν όλε οι χώρε μέλη τη Ένωση προσχωρούσαν στη σύμβαση του 1970, δεν θα προχωρούσαμε. Και πολύ σωστά έλεγε η κυρία ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα κεκτημένο το οποίο μπορεί να μα βοηθήσει για να οικοδομήσουμε κάτι, να προχωρήσουμε. Το να περιοριστούμε στο 70 για την επιστροφή, αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Ευχαριστώ. Monsieur... <laughs> Ευχαριστώ που μου δίνετε το, το λόγο και θα απαντήσω στην κυρία Βερζά στα Ιταλικά για να ξεφύγουμε από το, το πλαίσιο των γαλοφόνων. Εάν κατάλαβα καλά την ερώτηση αφορούσε μία αντίφαση στην παρουσίασή μου όταν αναφέρθηκα στο κριτήριο ή τα κριτήρια της επιμέλειας ως νέο κανόνα του ενιαίου δικαίου ή της ενοποίησης του δικαίου. Μιλώ λοιπόν για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού δικαίου, γι' αυτό και μίλησα για μια γενικότερη τάση που διαγράφεται. Σήμερα έχουμε ένα άρθρο 9 της οδηγίας όπου αναφέρεται ότι το βάρος της απόδειξης ορίζεται από το εθνικό δίκαιο. Δηλαδή η αρμοδιότητα αφορά ε, την κάθε εσωτερική ενόμη τάξη. Εάν λοιπόν αλλάξει τώρα το άρθρο 9 όπου διαγράφεται αυτή η αναφορά και όπου βλέπουμε ότι ο κάτοχος θα πρέπει να αποδείξει την επιμέλεια του και προσθεθούν και άλλα κριτήρια, τότε θα έχουμε ενιαία κριτήρια τα οποία θα αντικαθιστούν τη διαδικασία παραπομπής στο εθνικό δίκαιο. Αυτό δεν είναι πρότυπο αυτής της οδηγίας. Πριν αναφέρθηκα σε πολλούς κανονισμούς που είναι πιο δεσμευτικοί. Στον τομέα της ε, συνεργασίας στο νομικό και δικαιοδοτικό τομέα. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους κανονισμούς νέας γενεάς, δηλαδή μετά το 2005 5-6 τέτοιοι υπάρχουν όπου ο Ευρωπαίος νομοθέτης, δηλαδή τα τρία θεσμικά όργανα, ορίζουν προδιαγραφές ενοποίησης του κοινοτικού δικαίου. Άρα έχουμε κριτήρια τα οποία υποδεικνύονται, αλλά πρόκειται για ενιαία κριτήρια διότι έτσι και κατά αυτό το τρόπο διέπουν όλες τις εθνικές νομοθεσίες και δεν χρειάζεται η παραπομπή στον εθνικό δικαστή. Υπ' αυτή την έννοια μιλούσα για ενοποίηση. Δεν μιλούσα για ένα ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά για ε, ενία κριτήρια που να διέπουν τα κράτη-μέλη. Υπάρχει κάποιος από τους που θέλει να λάβει το λόγο. Κυρία. Ευχαριστώ. Απλώς θα ήθελα να διευκρινίσω το εξή σχετικά με το παράρτημα. Για την εξάλληψη του παραρτήματος είχα διατυπώσει αμφιβολίες σχετικά με το ότι αυτή η εξάλληψη ε, του παρατήρηματος ενισχύει την αποτελεσματικότητα της σύμβασης και ότι θα έπρεπε αυτό να θεωρήσουμε ότι είναι απόδειξη αναποτελεσματικότητας στην παρούσα κατάσταση της οδηγίας. Επικεντρωθήκαμε στους κινδύνους που θα δημιουργήσει η εξάλληψη του παρατήρηματος Απλώς ήθελα λίγο να εξηγήσω τις αμφιβολίες που υπάρχουν. Πιστεύουμε, ελπίζω να συμφωνούν και οι υπόλοιποι, πιστεύουμε ότι η εξάλληψη του παραρτήματος μπορεί να θεωρηθεί ως πρόοδος ε, στα πλαίσια του στόχου της οδηγίας. Ο στόχος είναι να καταπολεμήσουμε την παράνομη κυκλοφορία ε, των αγαθών του εθνικού πλούτου με στόχο την επιστροφή τους. Λοιπόν, το θέμα αυτό της αρχαιότητας μπορεί ε, να μας εμποδίσει στην πραγματοποίηση του στόχου μας. Αυτό είναι σημαντικό, διότι το αντικείμενό μας είναι αυτά τα αντικείμενα, σημαντικά αντικείμενα και βλέπουμε ότι οι μεγάλες συμβάσεις όπως είναι η Ντρουά δεν αναφέρεται στην αξία. Θα ήταν ίσως η ευκαιρία να προσεγγίσουμε την οδηγία από τις διεθνείς πράξεις. Επίσης η νομική ανασφάλεια μπορεί να προκύπτει από ε, την εκτίμησή μας ε, ενός πίνακα, ενός εργοτέχνης κτλ. Πάντα εδώ πέρα υπάρχει το θέμα της νομικής ασφάλειας ή ανασφάλειας. Επίσης πρέπει να υπάρχει αυτή η υποχρέωση της δέουσας επιμέλειας επειδή ορισμένα πολιτιστικά αγαθά δεν έχουν ε, εκτιμηθεί όπως τα θρησκευτικά αντικείμενα κτλ. Ορισμένε περιπτώσεις αναφέρεται η αξία τους και σε άλλες δεν αναφέρεται. Για όλους αυτούς τους λόγους Πιστεύω ότι η εξέλιξη του κειμένου είναι σωστή και το θέμα ότι δεν αναφέρεται το, η αξία τους και η αρχαιότητα μπορεί να θεωρηθεί ως πρόοδος. Τώρα, ε, η κατηγοριοποίηση, οι κατηγορίες. Ο Λιάρ Προσέ είπε ότι πρέπει να διατηρήσουμε τις κατηγορίες που είναι ένας καλός δείκτης Αυτές είναι ανοιχτέ κατηγορίες όμως. Δεν, ε, ο εθνικός πλούτος ε, περιλαμβάνεται, αλλά υπάρχει και η τελευταία κατηγορία που περιλαμβάνει τα πάντα, δηλαδή ε, κάθε είδους αντικείμενο το οποίο δεν ανήκει στις προηγούμενες κατηγορίες. Κύριε Μερσέ, νομίζω ότι ε, ως προς αυτά που μόλις είπε η κυρία Κορνού για το άρθρο υπαριθμών 1, το άρθρο αυτό μας απασχόλησε ιδιαίτερα ως κοιόδης ως προς τη διαγραφή του παραρτήματος, διότι συμμερίζουμε τις επιφυλάξεις που προανέφερε η συνάδελφος. Ε, κυρία Κορνού, με συγχωρείτε που σας το λέω έτσι ομά, αλλά η απάντησή σας δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Ως προς τη γραφή του παραρτήματος προβάλαμε το γεγονός ότι αντίθετα με τον τίτλο του, σε αντίθεση με τον τίτλο του, το κείμενο αυτό ε, ήταν πολύ δεσμευτικό για τα κράτη-μέλη. Και υπήρχε το θέμα του κατοφλίου ε, από χρηματοδοτικής πλευράς. Έτσι ε, πρέπει, τα ρίχνουμε όλα ε, στον Κεάδα Σιλίβδιν. Εάν το ε, θέμα είναι μεταξύ κατοφλίου και αρχαιότητας, τότε προτιμώ το κατόφλι. Και ας πούμε ότι το παράρτημα δεν πρέπει να είναι δεσμευτικό, αλλά ενδεικτικό. Και μην το διαγράψουμε. Γι' αυτό βρίσκω ότι οι απαντήσεις και οι συζητήσεις που έγιναν δεν είναι ικανοποιητικές διότι αν ο στόχος είναι να φτάσουμε προς την εναρμόνιση και όχι την ενιοποίηση έτσι ώστε η επιστροφή να είναι ε, ευκολότερη, τότε προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε. Γιατί οι επιστροφές ε, εδώ και 20 χρόνια, ο ρυθμός επιστροφών είναι δυσδιάκριτος, είναι κάτι το πολύ απογοητευτικό. Εάν ε, παραμείνουμε σε αυτό το γενικό πλαίσιο, με το νέο άρθρο υπαριθμών 1 δεν ε, ικανοποιούμαστε. Θα θέλαμε να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο, διότι αυτή τη στιγμή έχω πολλές αμφιβολίες και τις οποίες διατηρώ. Ευχαριστώ κύριε Πεζέ. Πρόκειται για ένα ε, εξαιρετικά νομικού χαρακτήρα ζήτημα που θα πρέπει εμείς να το προσεγγίσουμε από την πλευρά του, ε, πολιτιστικού περιεχομένου και όχι όσον αφορά τις ε, νομικές επιτυχίες. Νομίζω ότι περισσότεροι από εμά δεν είμαστε νομικοί, δεν είμαστε κατάλληλοι για να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Δικό μου το σφάλμα κυρία Μπεζέ, ε, γιατί νομίζω ότι σχεδόν σας ανάγκασα να καταρτήσετε αυτήν την ε, έκθεση. Σας ζητώ συγγνώμη εκ των υστέρων. Εγώ, είναι, μου είναι πολύ δύσκολο, δεν μπορώ να καταλάβω ε, ποια είναι η βελτίωση με την καινούργια πρόταση. Όταν τα ίδια τα έθνη μπορούν να αποφασίσουν τι είναι εθνικός θησαυρό για τα ίδια, τότε θα υπάρχουν μεγάλες διαφορές και ίσως ε, υπάρξει, δεν ξέρω αν από αυτή την διαδικασία μπορεί να προκύψει ε, μια δικαιότερη ρύθμιση του ζητήματος. Ε, το παράρτημα αυτό δίνει κάποιες ε, οδηγίες αφού κάθε έθνος μπορεί να αποφασίσει τι είναι ο εθνικός του θησαυρό. Και υπάρχει βεβαίως μια ε, επιθυμία προς ενιοποίηση και εναρμόνιση που δεν συνάδει απαραίτητα με την πυκλομορφία των πολιτισμών. Και αναρωτιέμαι, αν έχουμε την, αφού έχουμε την UNIDROIT, ε, γιατί δεν μπορούμε να πείσουμε και τις 28 χώρες μέλη να ε, επικυρώσουν αυτή τη σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειαζόμασταν καν οδηγία. Γιατί λοιπόν πρέπει να καταρτήσουμε οδηγία όταν θα μπορούσαμε να λύσουμε το ζήτημα μέσω της ε, σύμβασης. Εγώ στον πολιτικό τομέα είμαι πιο πολύ υπέρ των συμβάσεων παρά των οδηγιών. Νομίζω ότι ε, από αυτή την άποψη είναι κάπως αμφιλεγόμενο το ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει έχουμε την οδηγία. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είναι σκοπός όλων των κρατών μελών και οι 28 χώρες μέλη να επικυρώσουν την Ουνιντρουά. Διότι η Ουνιντρουά πηγαίνει παραπέρα από την οδηγία. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε σε ποιους τομείς η Ουνιντρουά ε, βαίνει παραπέρα από την οδηγία. Μπορείτε να μας το πείτε σε δύο-τρεις προτάσεις ή είναι πολύ δύσκολο αυτό που σας ζητάω. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα ήδη το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης UNITROA είναι πολύ ευρύτερο εφόσον καλύπτει και την κλοπή όσο και την παράνομη εξαγωγή. Εφόσον στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε το 1992 ήταν η εσωτερική κυκλοφορία. Δηλαδή ο αρχικός στόχο ε, ήταν ο ίδιος ένα, αλλά όχι, όχι ο αρχικό, στόχο ήταν διαφορετικός. Βεβαίω τα πράγματα εξελίχθηκαν από τότε. Η σύμβαση Unidroit, αν θέλετε, έχει το μειονέκτημα για ορισμένε χώρες, ότι αντίθετα από τη σύμβαση του 70, όπου σε ορισμένο βαθμό αυτά τα μέσα ε, είναι όχι άδεια κουτιά, αλλά μισογεμάτα κουτιά. Δηλαδή εξαρτάται από τι θα κάνουν με αυτά οι χώρες. Οι χώρες έχουν απόλυτη ελευθερία και είδαμε ότι αν ο στόχο είναι η επιστροφή των αγαθών, δεν πρέπει να αφήσουμε πολύ μεγάλη ελευθερία στα κράτη. Όχι επειδή δεν πρέπει να είναι ελεύθερα τα κράτη, αλλά επειδή η μη ομοιομορφία είναι αρνητική. Δεν φτάνουμε στο στόχο μας το βλέπουμε στη Σύμβαση του 70 εφόσον στράφηκαν σε εμά για να λύσουν τα πολύ σημαντικά προβλήματα και το ουσιαστικό πρόβλημα εδώ είναι η προστασία ε, στην περίπτωση καλής ε, πίστης θέμα το οποίο δεν ελύθηκε το 70, εν μέρη λύεται μέσα από την οδηγία, αλλά το βάρος απόδειξης που δεν είναι στον κάτω αυτή τη στιγμή διαιωνίζει το πρόβλημα. Δεν σας κρύβω ότι ο δισταγμός όσον αφορά τη σύμβαση Ινιδρουά ε, ε, είναι διπλός είτε όσον αφορά ανοιχτά την αγορά τέχνης και εδώ πρέπει να πω ότι από τότε που υιοθετήθηκε η σύμβαση Unidroit πολλές χώρες της αγοράς τέχνης ε, που δεν είχαν ακόμα προσχωρήσει τη σύμβαση του 70 της UNESCO προσχώρησαν και η πιο επιμελής θα έλεγα στην εθνική τους νομοθεσία εφαρμογής αυτής της σύμβασης περιέλαβαν ορισμένα στοιχεία της Γιουλιντρουά και κυρίως ε, την δέουσα επιμέλεια. Γνωρίζουμε, τουλάχιστον στην Ελβετία, για να αναφέρω μια χώρα που δεν ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζουμε ότι αυτές οι νέες διατάξεις σε τίποτα δεν παρεμπόδισαν το παράνομο εμπόριο. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, η αγορά τέχνης τον αναγνωρίζει, δεν υπήρχαν νομικές ε, ε, ε, αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά τέχνης. Το αντίθετο, θα έλεγα ότι υπάρχει μια γενική αναγνώριση για, αυτούς τους, για αυτή την αγορά. Τώρα, άλλη αντίδραση άλλων χωρών είναι νομικής μορφής και το είδαμε στα σχόλια που έγιναν για την αναδιατύπωση τη οδηγία. Ορισμένοι είπαν ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε, διότι αυτό δεν συμβαδίζει με το δικό μα το νόμο, την νομοθεσία μα. Ναι, συμφωνώ, αλλά εάν οι διεθνεί πράξει, περιφερειακές, η διεθνή νομοθεσία, περιφερειακή, η διεθνή, ε, ανικατοπτρίζει την εθνική νομοθεσία, τότε δεν θα είχαμε τίποτα παραπάνω. Πρέπει να προχωρήσουμε, η κυρία Βερζέ το είπε, πρέπει κάπως να προχωρήσουμε. Έχουμε μία βάση και πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να συμφωνήσουμε ω προ το στόχο. Τι θέλουμε. Περισσότερε επιστροφέ, αγαθών, μεγαλύτερη προστασία. Πρέπει να συμφωνήσουμε. Και αυτό ήταν στη βάση των διαπραγματεύσεων της UNIDROIT. Ορισμένα ε, δικαιώματα είναι θεμελιώδη, αλλά ο στόχος μας πρέπει να είναι να διευκολύνουμε την επιστροφή των αγαθών. Και τι πρέπει να κάνουμε. Το γαλλικό δίκαιο είναι ένα δίκαιο το οποίο φυσικά ε, είναι νομικής μορφής, αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένες πράξεις. Εδώ και καιρό τα πολιτιστικά αγαθά αναγνωρίζονται ως ανήκοντα σε μια κατηγορία που θα πρέπει να διέπεται από ειδικού κανόνε. Μπορούμε να το λέμε, αλλά εδώ έχουμε και την δυνατότητα να το αποδείξουμε. Εάν τα πολιτικά αγαθά είναι πράγματι τόσο σημαντικά ώστε θα πρέπει να την χάνουν προστασίες, τότε θα πρέπει να ε, την χάνουν παρεκκλήσεων από, το, από τη Γενική Νομοθεσία. Συνεπώ, ε, τα επιχειρήματα τη μη συμβατότητα με το Εθνικό Δίκαιο και άλλωστε οι περισσότερε χώρε που δεν προσχώρησαν στην Ιντρουά είπαν ότι Τίποτα στη σύμβαση δεν είναι ασυμβίβαστο με το δίκαιό μας. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης και σκοπιμότητας. Ναι, κύριε Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι ως προς το ερώτημά σας. Εάν κατάλαβα καλά, μας λέτε ότι υπάρχουν ε, κατά βάθο δύο ε, διεθνείς συμβάσεις και ίσως θα επαρκούσαν. Στην πραγματικότητα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αντίθετη πλευρά, δηλαδή ότι η οδηγία υπάρχει, προϋπάρχει, όπως υπενθυμίσατε, αλλά δεν λειτουργεί πολύ καλά. Και ανακύπτει ότι οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών ε, εκφράστηκαν υπέρ μιας τροποποίησης ε, της οδηγίας για να λειτουργήσει καλύτερα. Βασίζεται στο άρθρο 114 της ε, λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Άρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει αυτή τη στην αρμοδιότητα. Απλώς θα πρέπει να βελτιώσουμε τους ε, μηχανισμούς αυτούς που προϋπάρχουν, της οδηγίας δηλαδή, και που κατέδειξαν ε, ορισμένες αρνητικές πλευρές. Τώρα κατανοώ την αντίρρηση της κυρίας Βερζιά, διότι μιλάμε για την επίτευξη μιας εναρμόνισης ε, των εθνικών νομοθεσιών. Αυτό μπορεί να γίνει με βάση ενιαία κριτήρια. Δηλαδή δεν επιβάλλουμε κάτι στα κράτη-μέλη, αλλά ορίζουμε ενοποιημένα κριτήρια έτσι ώστε να υπάρξει μια σύμπνοια στα κράτη. Και έτσι η συμπεριφορά θα είναι ίδια από τους εθνικούς δικαστές όταν αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο αίτημα επιστροφής με βάση την οδηγία. Ευχαριστώ. C'est euh, correct ou non C'est français, hein Cornu Oui. Bon, d'accord, allez-y. <laughs> Merci. Ευχαριστώ. Euh, Και εγώ θα ήθελα να πω επίσης ότι η οδηγία, αν πάμε πίσω, τη στιγμή που υιοθετήθηκε, είναι ένα μέσο, μια πράξη που αντισταθμίζει ε, η καλύπτη τα κενά προστασίας μιας ενιαίας αγοράς. Δεν πρέπει να το λησμονήσουμε αυτό, διότι τα συστήματα προστασίας των χωρών εξασθένησαν από την εξάλληψη των συνόρων, των ελέγχων στα σύνορα δηλαδή. Αυτό είναι το πνεύμα του κανονισμού και του ελέγχου απέναντι στις τρίτες χώρες. Και αυτή είναι η φιλοσοφία του συστήματος της οδηγίας. Αν ε, δεν υπάρχει πια αυτός ο μηχανισμός, τότε θα υπάρξει κίνδυνο όσον αφορά την προστασία του εθνικού πλούτου. Επίσης, λέτε γιατί δεν καταλαβαίνετε, γιατί θα παραπέμψουμε στις διάφορες χώρες τον ορισμό του εθνικού πλούτου. Αυτό υπάρχει, δεν δημιουργεί πρόβλημα. Το άρθρο 36 της συνθήκης το αναφέρει. Και λειτουργεί πολύ καλά. Δηλαδή τα κράτη-μέλη επιβάλλουν τους περιορισμούς τους όσον αφορά ε, τον έλεγχο ε, ή την απαγόρευση ε, της κυκλοφορίας, ε, των ε, πολιτιστικών αγαθών και των έργων τέχνης. Και αυτό το άρθρο ζητεί από τα κράτη-μέλη να προσδιορίσουν τον εθνικό τους πλούτο. Συνεπώς είμαστε συμβατοί με αυτό το άρθρο και δεν υπάρχει πρόβλημα. Κυρία Σνάιντερ ξέχασα να πω τα εξή τα συμπεράσματά μου. Νομίζω ότι η αναδιατύπωση της οδηγίας είναι ύψης της ε, σημασίας μέσα στα πλαίσια της ε, τελικής ε, κύρωσης, διότι η οδηγία θα πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Εάν η αναδιατύπωση ε, ξαναλάβει υπόψη στοιχεία όπως την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης ή το θέμα της επιμέλειας σημαίνει ότι κινούμαστε προς τα εμπρός. Θα ήταν κάτι το θετικό γιατί τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να προβάλλουν επιχειρήματα για να μην κυρώσουν Εάν τους αφήσουμε λοιπόν την ελευθερία κύρωσης ή μη, τότε θα τηρήσουν στάση επιφύλαξης και θα δεχτούν τις πιέσεις από συγκεκριμένα ε, λόμπι. Εάν όμως υπάρχει αυτή η θετική προσέγγιση, εφαρμοστεί αυτό το θετικό δίκαιο, θα έχει ε, σοβαρές θετικές επιπτώσεις. Λοιπόν, ε, θεσπίζουμε νόμους που ονομάζονται οδηγίες Πρόκειται δηλαδή για νόμους πλαίσια που μεταφέρονται στις εθνικές νομοθεσίες. Αυτό δεν αφορά, μια τέτοια υποχρέωση δεν αφορά τη σύμβαση. Μπορεί μια σύμβαση να ε, ε, εφαρμοστεί και διαφορετικά. Αυτή είναι η διαφορά μας και με το Συμβούλιο. Το καταλάβαμε αυτό. Αυτό που θέλαμε να μάθουμε είναι ποιες είναι οι μεγάλες ε, διαφορές μεταξύ UNIDROIT και ε, της οδηγίας. Τώρα, η κυρία Παζιά ε, είχε καθήκον να εξαγάγει κάποιο συμπέρασμα. Ε, δεν πρέπει να το κάνει τώρα, μπορεί να το κάνει μαζί με την υποβολή της εισήγησής της και μπορούμε βεβαίως και να μαλώσουμε σε μια επόμενη φάση. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, μίλησαν, διότι οι παρεμβάσεις τους ήταν ποιοτικέ και επιτρέπουν ε, να δώσουμε φως σε μια δύσκολη νομική συζήτηση. Νομίζω και για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας κυρία Πρόεδρε, αυτό το οποίο βρίσκεται πίσω από όλα αυτά είναι η προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Αυτό το ονομάζουμε την πολιτιστική εξαίρεση. Εάν το άρθρο 36 υπάρχει στις συνθήκες, εάν η οδηγία του 93 εφαρμόστηκε, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει πολιτιστική εξαίρεση. Και δεν θέλουμε και συμφωνούμε φαντάζομαι σε αυτήν την Επιτροπή τουλάχιστον δεν θα θέλαμε τα πολιτιστικά αγαθά να αντιμετωπίζονται ως κοινά αγαθά. Λυπούμε όμως επειδή εξετάζουμε αυτό το θέμα μέσω του θέματος της αγοράς. Επειδή η νομική βάση είναι το άνοιγμα της αγοράς στην αρχή της δεκαετίας των 90. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν είμαστε στριμωγμένοι, βρισκόμαστε μπλεγμένοι μέσα σε αυτό το νομικό πλαίσιο. Αλλά δεν θέλω να αμφισβητήσω και πάλι αυτό το νομικό πλαίσιο και ε, δεν θα ήθελα να προτείνω ούτε την ε, τροποποίηση του άρθρου 36. Ε, αυτό είναι αντίθετο με τα όσα συνηθίζω. Μέχρι την πέμπτη μεσημέρι πρέπει να συντάξω ρεσμένα πράγματα εάν θέλουν οι μεν και οι δεν να έχουν ένα έγγραφο μεταφρασμένο μέσα στα προβλεπόμενα περιθώρια. Θα πρέπει λοιπόν να περιλάβουμε ορισμένα πράγματα στις σκέψεις, διότι το πλαίσιο της αναδιατύπωσης οδηγίας είναι περιορισμένο, επειδή πρόκειται για αναδιατύπωση. Δεν έχουμε πολύ μεγάλα περιθώρια λιγμών. Νομίζω όμως, αν κατάλαβα καλά τουλάχιστον τη θέση του Συμβουλίου, έχουμε κάποια περιθώρια λιγμών εδώ, θα μπορούσαμε να περάσουμε με ένα μηνύματα υπό με την έννοια που θέλουμε να δώσουμε σε αυτό το θέμα για να διευρύνουμε αυτή την οδηγία σε σχέση με τα όσα διακυβεύονται. Το ουσιαστικό, θα τα πω στο νου μου, είναι το πρώτο άρθρο, γιατί μπορεί να ασφάλω, αλλά νομίζω ότι τα κράτη-μέλη κάπως προχώρησαν εδώ και θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια συνένεση, σε μια συμφωνία ως προς τη σύνταξη του πρώτου άρθρου. Υπό τον όρο ότι εμείς οι ίδιοι δεν θα κάνουμε αυτό που κάνει η Κομισιόν. Ανάμεσα δηλαδή στις δύο έννοιες, να το ξεκαθαρίσουμε. Να ξεκαθαρίσουμε στις δύο έννοιες, δηλαδή την ε, καλή πίστη και τη δέουσα επιμέλεια. Για το πρώτο άρθρο δεν έχω ακόμα ξεκαθαρίσει τις σκέψεις μου. Ε, ε, και άλλωστε θα δω την Τετάρτη το πρωί τους και όλους τους για να το δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες. Ήταν πολύ διαφωτιστικά τα όσα μας είπαν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Επομένως κλείνουμε το εργαστήριο και μπορώ να παρακαλέσω να αποχωρήσουν όλοι όσοι δεν ανήκουν στους συντονιστές. Εσείς μπορείτε να μείνετε αν θέλετε.